Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Αν δεν έχουμε άλλο σχολείο μπορούμε να πάμε στο σημείο 7 τη διατάξεω. Την υλοποίηση της ετήσιας, μάλλον της κοινή πολιτικής ε, ε, ασφάλειας, ε, εξωτερικής και πολιτικής ασφάλειας, της ΚΕΠΑ, εν πάση η ετήσια έκθεση να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους αυτούς που συνεισέφεραν στο, στη σύνταξη του κειμένου και ιδιαίτερα τους Σκιώδης. Λάβαμε 398 τροπολογίες στην αρχικό σχέδιο ετησίας εκθέσεως. Τροπολογίες που εξέφρασαν υποστήριξη στη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την προστασία του, της πολυμέρειας μέσω μιας πιο γεωπολιτικά σημαντικής τάσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολλοί από εσά είπατε ότι προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματικός παγκόσμιο παίκτη, θα πρέπει να έχουμε να ενισχύσουμε τα μέσα που έχουμε διάθεσή μα και να είμαστε πιο συνεπεί στη στάση μας. Επίση, αρκετέ τροπολογίες σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΑ Επίση αρκετέ τροπολογίε για την ε, πολιτική γειτονία, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το μελλοντικό ρόλο του ΝΑΤΟ. Αρκετοί αναφερθήκατε και σε αναδυόμενες οικονομικέ δυνάμει στην Ανατολική Ασία και τι απειλέ που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για την κυβερνασφάλεια, υβριδικέ απειλέ και κλιματική αλλαγή. Προσπαθούμε τώρα να συνδυάσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες για να έχουμε μια συνεπή έκθεση και υπολογίζω στην επικοδομητική συνεργασία με τους Σκιώδης. Επόμενη συνάντηση με τους οποίους θα έχουμε στο Στρασβούργο 28 Νοεμβρίου. Να ακούσω λοιπόν τώρα τις απόψεις σας για τις 398 τροπολογίες. Ο κύριος Λόπεθ αρχικά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Τσάβη, ευχαριστώ πρόεδρε εμείς Χωρί να πάω σε λεπτομέρειε τώρα των 400 σχεδόν αυτών τροπολογιών, θέλαμε να πούμε πρώτον να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή μας και πρόεδρο για τη δουλειά. Είναι ένα πολύ καλό σημείο κίνησης διαπραγμάτευση Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια καλή έκθεση και συνεντική. Τέσσερα τώρα στοιχεία που θέλαμε να περάσουμε με τις τροπολογίες μας να ενισχύσουμε τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ασφάλειας και της ειρήνης, να είναι δηλαδή ένας ισχυρός φορέας, παίκτη και να στηρίζεται στα μέσα της την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, διπλωματία με συγχωρείτε, την ΚΕΠΑ και τον ε, είπα το εκπρόσωπο και βεβαίως την ε, δουλειά που κάνει ήδη το Κοινοβούλιο. Να υπογραμμίσουμε βέβαιως επίσης τις αρχές που διέπουν την εξωτερική μας πολιτική. Το αρχικό κείμενο είχε πολλές και διάφορες παραπομπές και συμφωνούμε για ένα παγκόσμιο σύστημα ε, πολυμέρειας υποκανόνες. Ένα πλαίσιο κανόνων και ένα πλαίσιο πολυμέρειας που υφίστανται απειλές σήμερα. Εμείς θέλαμε Κάτι ακόμα συνεισφέρουμε για την θεματολόγιο 2030, τη Συμφωνία του Παρισίου, το μέλλον του ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες ε, ασφάλειας και ειρήνευσης. Επίσης, τις απειλές, ε, τις πολύ περίπλοκες που αντιμετωπίζουμε πλέον τις υβριδικές, με νέα φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή, την ανισότητα, ε, τις ψηφιακές απειλές, γενικώ στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία και έναντι αναδειωμένων νέων δυνάμεων πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και τέταρτον, αναφερόμαστε σε κάποια ίσως περιφερειακής φύσεως ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό, στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ δηλαδή την εδαφική συνοχή και την κυριαρχία με τους, γειτονικούς, με τους ανατολικούς μας γείτονες, την συνεργασία με τις χώρες του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και μια συνεργασία με την ε, Νότιο Αμερική περιοχή που γνωρίζει μεγάλες ε, αναταράξεις αυτή τη στιγμή. Συνολικά όμως πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση συμβάλλει στη δουλειά του Κοινοβουλίου για την κοινή διαμόρφωση τη ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Thank you. Shabby Lopez, looking forward to Thursday morning. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόπες. Θα τα ξαναπούμε το, την Πέμπτη το πρωί στο Στρασβούργο. Κυρία Βάουτμανς για το Ρινιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Συγητά. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Έχει πολλά θετικά στοιχεία η έκθεση που μας υποβάλλεται. Είναι πολύ σημαντικότερο που θα έχουμε και μια καινούργια επιτροπή να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου για, την, για τα θέματα αυτά, να πούμε ποια είναι ε, στοιχεία αυτής της πολιτικής που τα θεωρούμε σωστά και τι πρέπει να αλλάξει. Στην έκθεση αναφέρονται πολλά από αυτά. Εμείς έχουμε βάλει τροπολογίε που πηγαίνουν προ την εξή κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερη ενότητα, τόσο, όλο και περισσότερη αλληλεγγύη, έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική για τα θέματα αυτά. Δεύτερον, αυτό δεν μπορεί να συμβεί και να είμαστε ενωμένοι και να φαινόμαστε ενωμένοι προς τα έξω εάν δεν έχουμε μια ε, ουσιαστική εφαρμογή των ιδίων αξιών και στο εσωτερικό. Τρίτον, δεν αρκεί πλέον η ήπια δύναμη, το soft power, αλλά επίσης και μια ουσιαστική ε, δύναμη ε, που να μπορεί να επιβάλλει την, ε, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αυτό σημαίνει ότι βεβαίως θα αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να λειτουργεί και προλαμβάνοντας καταστάσεις αλλά και ανταποκρινόμενοι σε αυτές. Επίση, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια καλύτερη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα των πόλων, του Βορείου και του Νοτιού Πόλου, τη χρήση του. Και επίση, θα πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ο, κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζεται πια αυτή η σχέση, κάποιοι λένε ότι ο καθένας μπορεί να λύσει τα προβλήματα μόνος του. γιατί εμάς, εμείς πιστεύουμε ότι είναι και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική η σχέση με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε Χίλτα Ζερόμ Λεβιέρ για το ID. Σας ευχαριστώ. Δεν θα εκπλαγείτε από τη θέση που θα λάβω. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα πρέπει να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό επίπεδο και α, ποιότητα μάλλον της έκθεση που μας υποβάλατε. Εμείς ως ομάδα πολιτική γενικά πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις αρμοδιότητες τους. Με βάση τις συνθήκες και εφαρμόζεται μόνο εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση από όλα τα κράτη-μέλη. Σε καμία περίπτωση, αν σεβόμαστε τη δημοκρατία, δεν μπορούμε να, δεχτούμε ε, παρεμβάσεις στην εθνική καριερχία των κρατών. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην έκθεσή σα προτείνετε να πάμε όλο και περισσότερο προς μια ομοσπονδιοποίηση τη εξωτερική πολιτική τη Ένωση και όλο και περισσότερο να λαμβάνονται αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία. Εμεί δεν το επιθυμούμε. Επιθυμούμε να υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών, μεταξύ εθνικά ανεξάρτητων κρατών μελών, ε, προ την επίτευξη κοινών πολιτικών. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν δεχόμαστε και αυτό τον όρο που εισάγεται για την ε, αυτόνομη ε, στρατηγική ε, τα αυτόνομα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύουμε ότι μας πάει προς περισσότερη ομοσπονδιοποίηση. Γνωρίζουμε ότι πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε στον κανόνα της ομοφωνίας, ιδιαίτερα αυτό ισχύει σε ζητήματα στρατηγικά ή διπλωματικά. Υπάρχει πρόταση να γίνει όλο και πιο αυτόνομη η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της, ε, της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας, όμως εμείς θέλουμε αυτό όλο να, να, να διευκρινίζεται ότι θα γίνεται επί τη βάση της αρχής της ομοφωνίας. Εμείς πιστεύουμε επίσης ότι είναι η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ όλο και ακόμα ε, δεν είναι ε, δεν συνεχίζει να είναι μάλλον απαραίτητη, δεν θεωρούμε ότι η αυτόνομη ε, συνεργασία, η αυτόνομη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν το στρατηγικό ε, σκέλος του ΝΑΤΟ. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να χάσουν την δικιά τους δικαίωμα ή τη δυνατότητα παρέμβασης για τα στρατηγικά τους συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ζερόμ, για το ECR, η κυρία Φατίκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Σίγητα να σας συγχαρώ για το έργο σας μέχρι τώρα. Περιμένω με αγωνία να δω πώς θα διαμορφωθούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς το τελικό κείμενο της θετήσης έκθεσης για την ΚΕΠΑ, ιδιαίτερα σε ταραγμένες περιόδους όπως αυτή. Παρ' όλα αυτά, ε, εγώ έχω ε, την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε όταν χρειάστηκε να γίνει η ακρόαση του είπα του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλεια και καταφέραμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις εκεί. Επίσης τα θέματα αυτά θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ιδιαίτερα και σε σχέση με τους πόρους που θα χρειαστούν. Ευελπιστώ λοιπόν ότι και με εντατική εργασία στο Στρασβούργο θα καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις και σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε Άννα. Κανένας από την ε, Γκουε, όλη η ομάδα είναι στη Φιλανδία από ό,τι ε, γνωρίζω. Ε, περνάμε στο EPP. ο κύριος ε, Σικόρσκι. Ελπίζω και εσείς ε, για την, την Washington ε, να εκπλαγεί κατά όσο και εγώ. διότι με όλες τις διαφορές που έχουν οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκράτες μεταξύ τους συμφωνούν στο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες βρίσκεται σε μια ε, παγκόσμια ε, αντιπαλότητα για κυριαρχία με την ε, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και, προς, και αυτή η αντιπαράθεση έχει βρίσκει υποστήριξη και στα δύο κόμματα. Ε, υπάρχουν προσπάθειες να μας πείσουν ε, για μια ε, κοινή θέση προς την Κίνα κάτι το, μια διαδικασία την οποία κάνανε πολλές φορές στο παρελθόν όμως η, κοινωνία η Κίνα είναι πολύ πιο σημαντική όταν σκεφτόμαστε την τρέχουσα κυβέρνηση και το στυλ που έχει έχει κάποια δίκαια, ότι έχουν, ε, γίνεται κατάχρηση του ε, εμπορικού συστήματος, ότι ορισμένες ε, διαδικασίες οι οποίες έχουν εμπορική φύση, στην πραγματικότητα είναι, έχουν στρατηγική φύση. Για παράδειγμα έχουμε την τεχνολογία η οποία κλέβεται από ξένες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να το επιβραδύνουμε. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας προτείνω αλλά και να ε, ζητήσω την υποστήριξή σας ε, για τις ε, ε, τροπολογίες μου 137 ε, και 357 όπου προτείνω να έχουμε ένα εθελοντικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων μεταφορών τεχνολογιών στις χώρες που μας απασχολούν και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι ε, οι ανταγωνιστές ε, δεν θα έχουν ε, ένα άδικο πλεονέκτημα εις βάρος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να ενσωματώσω την τροπολογία σας, όμως θα πρέπει να έχω και την υποστήριξη των σκιωδών. Είμαι αισιόδοξο παρόλα αυτά. Ο κ. Παζέσκου τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να σας ε, συγχαρώ ε, και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για την έκθεση αυτή. Έχω υποβάλει αρκετές ε, τροπολογίες, όμως οι τροπολογίες αυτές Ε, έχουν ως ε, στόχο τους ε, να υπάρξει περισσότερη αυστηρότητα αλλά και διάβγεια στην κοινή εξωτερική πολιτική μας το οποίο θα πρέπει να είναι και το βασικό μήνυμα της έκθεσης αυτής, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει η στρατηγική αυτονομία την οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο έχουμε μια κατακαιρματισμένη εξωτερική πολιτική, τότε ε, τόσο λιγότερο θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις ε, παγκόσμιες αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο και πιστεύω ότι μια ενιαία εξωτερική πολιτική και ε, μια συμφιλίωση με τους συμμάχους μας αλλά και η δημιουργία νέων συμμαχιών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηριχθεί. και η ιδέα της σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με τους διατλαντικούς μας εταίρους, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ύστερα από τη, ακούγοντας τις δηλώσεις διαφόρων ε, ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γι' αυτό το λόγο εκτιμώ ε, το ότι υπάρχει αυτή η πρόταση για μια ενίσχυση των σχέσεών μας και κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνω και στις τροπολογίες μου εάν ε, συνεχίσουμε ε, κάποια ε, χρόνια ακόμα με αυτή την κατακαιρματισμένη εξωτερική πολιτική, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει λιγότερο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο και εν τέλει θα γίνουμε λήπτης πολιτικών στρατηγικών από Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείες με αποτέλεσμα να πρέπει να ε, βιώνουμε τις ε, συνέπειες. Ε, θα μπορούμε μονάχα να αντιδρούμε αντί να δρούμε στα φόρα όπου λαμβάνονται οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και από το ECR Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την ε, ε, πολύ καλά συνταγμένη έκθεσή σας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία από ρεαλιστικής άποψης δεν είναι αρκετά. Ε, διότι ε, δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι οι εξωτερικές ε, σχέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των ανεξάρτητων κρατών. Και γι' αυτόν τον λόγο εμείς από το ECR έχουμε ε, υποβάλει μία γνωμοδότηση. Μην αναφέρομαι ε, στην πρότασή σας ε, για την κατάργηση του δικαιώματος ανησυχηρίας στο Συμβούλιο και αυτού θα πρέπει να υπάρχει ε, πλειοψηφία. Λέτε ότι ο λόγος είναι η αποτελεσματικότητα, όμως εδώ βλέπω ότι κινούμαστε προς την κεντροποίηση. Ε, οι πρωτεύουσες των κρατών μελών έχουν τις ε, δικές τους εξωτερικές πολιτικές. Ε, αυτό είναι, προς, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εθνικών συμφερόντων και γι' αυτό το λόγο καλό την πλειοψηφία αυτής εδώ της Επιτροπής να το ξανασκεφτούμε το θέμα αυτό. Δεν θεωρούμε ότι ε, αυτό ε, μπορεί να επιτευχθεί έτσι όπως ε, το παρουσιάζει η συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Η εξωτερική πολιτική λοιπόν συνδέεται άμεσα με την έννοια της ε, ανεξαρτησίας των κρατών, οπότε εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή τη θέση. Ωραία συνάδελφοι, σας ευχαριστώ συνάδελφοι. 28 Νοεμβρίου θα συζητήσουμε στο Στρασβούργο και ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε όσες περισσότερες τοπολογίες μπορέσουμε. 4 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ψήφο στην ΑΦΕΤ. 13 με 16 Δεκεμβρίου θα πάει στην Ολομέλεια. Τώρα εγώ καλούμε να λάβω το λόγο πλέον για την έκθεση ε, καθότι ο κύριος Ντανζό ζητώντα συγγνώμη που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του θα διαβάσω λοιπόν αυτά που έχει να μας πει. Ζητάει συγγνώμη ο κύριος Ντανζό που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Παρουσίασε την ετήσια έκθεση πριν από δύο εβδομάδες στην Επιτροπή της ε, CSTP οι ομάδες ε, τοποθετήθηκαν. Συνολικά 500 ε, τροπολογίες έχουν υποβληθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Η δουλειά της μετάφρασης των τροπολογιών ακόμα συνεχίζεται. Θα είναι διαθέσιμες μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Και κατόπιν ο κύριος Ντονζόν θα διατρέξει όλες τις τροπολογίες και θα συζητήσει το συντομότερο δυνατόν με τους κοιόδης στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα και όποιο σχόλιο αναφερθεί σήμερα θα του διαβιβαστεί. Ο κ. Τονζό θα έχει, ελπίζει να έχει μια επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδεις για να έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο. 4 Δεκεμβρίου στην ΑΦΕΤ και τον Ιανουάριο του 20 στην Ολομέλεια. Του Αγνώ, λοιπόν, η δικιά μου έκθεση είναι το, το Δεκέμβριο, του Αγνώ πάει για τον Ιανουάριο και οι δύο το Δεκέμβριο. Η δικιά μου η έκθεση υποτίθεται ότι θα, βο... θα ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Του, του κυρίου Ντονζόν θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο, συνήθως δεν πάνε μαζί. Okay, well, we'll figure that out in the meantime. Colleagues, this was Mr. Dajon's statement. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς έχουν ε, τα χρονοδιαγράμματα. Αυτά για την έκθεση του κ. Τονζό, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Κομπίλιος. Ένα σύντομο σχόλιο, Πρόεδρε. Ε, έχουμε πολύ καλές ιδέες στην έκθεση αυτή. Αυτό που εγώ θα πρότεινα παρά το γεγονός ότι εμείς προτείναμε κάποια, κάποιες από αυτές τις κοινέ τροπολογίες. Υπάρχει ένα ζήτημα που απαιτεί μια κάποια σαφήνεια. Η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας που ακούγεται όλο και περισσότερο. Δεν είμαστε ενάντι, αλλά χρειαζόμαστε μια σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούμε με την έννοια αυτή. Δηλαδή πού χρειαζόμαστε στη στρατηγική αυτονομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πού για το ΝΑΤΟ. Αυτό λείπει από την έκθεση. Μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι μιλούμε για ευχές εδώ, ευχολόγιο που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Τι εννοούμε με τη στρατηγική αυτονομία, μιλούμε τα πυρηνικά όπλα ή κάτι άλλο. Γιατί σε πέρα, γιατί πέραν αυτό το, το, το, ΝΑΤΟ είναι το πλαίσιο της αποτρεπτικής μας ικανότητος εναντί επιθετικών ε, τρίτων χωρών όπως η Ρωσία. Ιδάλλως, ποιος είναι ο ρόλος της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και πώς θα τη χρησιμοποιούσαμε. Θα εκτιμούσα να υπάρχει μια τέτοια έτσι, διευκρίνηση. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Στο μεταξύ να σας πω ότι και οι δύο εκθέσεις θα πάνε στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. και ζητώ συγγνώμη επίσης που έδωσα πρώτο το λόγο στον κύριο Καμπίλιο γιατί κανονικά ξεκινούμε με τους Σκιώδη. Αυτό το έκανε επειδή έλειπε ο Αγανό, αλλά τέλος πάντων. Ε, ο κύριος ε, Ρακόβαξ θα μιλήσω ογκρικά πρόεδρε ε, εκ μέρους των S&D καθότι είμαι σκιώδης εισηγητής για την έκθεση αυτή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και Άμυνες Υποβάλαμε ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε στενή και φιλικότατη συνεργασία με τον κύριο Ντονζό, τον οποίο ευχαριστήσαμε ήδη για τη συνεργασία. Τέσσερις σύντομες παρατηρήσεις, εφόσον μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. <clears throat> Πρώτον, σε καιρού που αντιμετωπίζουμε τόσες πολλές προκλήσεις και προβλήματα είναι ακόμα πιο σημαντικό να στοχεύουμε σε ακόμα μεγαλύτερη εναρμόνιση των εξωτερικών δράσεων μας της και παλαιοπολιτικής. Ο ομιλητής με Για τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης να μην ξεχνούμε ότι ο 20ος αιώνας ξεκίνησε με, μια, με ένα τραγικό πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια περιοχή που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα και εθνοτικές αντιπαραθέσεις με μεγάλη παράδοση και ιστορία. Είναι σημαντικό να προσέχουμε την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων λοιπόν. Τρίτον, μιλήσαμε πρόσφατα για τις υβριδικές απειλές. σε εκθέσεις άμυνας πρέπει να αφιερώνουμε πάντοτε πιστεύω διακριτό κεφάλαιο στις βρυδικές απειλές. Και τέταρτον, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχαμε ειδική πλειοψηφία σε θέματα ασφαλείας και άμυνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής δεν είναι παρόν για τους Ρινιού. Άρα, Jérôme Rivière, ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αντίστοιχο πνεύμα με την προηγούμενη παρέμβαση, με αντίστοιχη προσέγγιση υποβάλλουμε τροπολογίες προκειμένου να εγγυόμεθα την ε, ανεξαρτησία και κυριαρχία των κρατών μελών στα θέματα πολιτικής ε, άμυνας. Δηλαδή οι στρατιωτικές ικανότητες σχεδιασμού ε, και αποτρεπτικές δυνάμεις αν θέλετε και η οργάνωσή τους στην ουσία αποτελούν μια απόπειρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέλθει στα θέματα κυριαρχίας των κρατών μελών και αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν πλαίσια συνεργασία πολύ επιτυχού ε, όπως η Airbus, ε, τα οποία σήμερα δεν θα μπορούσαν να λάβουν χώρα ε, υπό το πλαίσιο αυτό που έχουμε, όπου πνίγεται η ελεύθερη ε, πρωτοβουλία των κρατών μελών από τους πολλαπλούς κανόνες και διατάξεις και ρυθμιστικό πλαίσιο που επιβάλλει η Επιτροπή. Θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι είναι απολύτως κυρίαρχα τα κράτη-μέλη στις ε, στρατηγικές τους ε, επιλογές, ιδιαίτερα στους εξοπλισμούς. Και όπως έγραψε ο Αλμπέρ Καμού, είναι το να αναφερόμαστε εσφαλμένα στα πράγματα είναι το να περιγράφουμε λανθασμένα τον κόσμο. Και να δίνουμε κακό όνομα σε ορισμένες έννοιες. Ε, πολύ μιλούμε τελευταία για την Τουρκία. Εμείς θεωρούμε ότι τα, τα θέματα της συνεργασίας αυτής δεν θα έπρεπε να στρέφονται μόνο σε στρατηγικά ή δηλαδή πολεμικής ε, υλοποίησης θέματα, ε, καθαρά στρατιωτικής υλοποίηση θέματα, αλλά θέματα διαχείρισης, ε, πλαίσιο διαχείριση για τους ε, δορυφόρους, μεταξύ άλλων για τη διαστημική πολιτική. Ε, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να σα πείσουμε τέλο πάντων για το εύλογο των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ριβιέρ. Να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πίσω μέρος της αίθουσας να καλωσορίσουμε την διαθρησιακή ε, αντιπροσωπεία από τη Γεωργία που εκπροσωπούν τις Ορθόδοξες Μουσουλμανικές ε, αρ, ε, Αρμένικες κοινότητες της χώρας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερους για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζω να ε, έχετε μια παραγωγική επισκέψη στις Βρυξέλλες και επίσης να εκφράσω την ε, εκτίμηση της Επιτροπής μας, τις προσπάθειες που κάνετε ε, για την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή σας. Έχετε, έρχεστε από μια χώρα με μεγάλη ιστορία που εκπροσωπείται και από άξιους εκπροσώπους εδώ στο Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κύριο Κάλε Επίσης, φίλο της Γεωργίας, αν και δεν είναι το θέμα μας τώρα εδώ, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους προκεσκυκλισμένους μας και εγώ, λέει ο κύριος Γκάλερ. Για δέκα χρόνια ήμουν συντονιστής του ΕΛΚ για την κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλειας και με αυτή την ιδιότητα έχω υποβάλει και εγώ κάποιες τροπολογίες στην έκθεση που θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν υποκοδομητικά. Εγώ θέλω να επανέλθω σε ένα ζήτημα που αναφέρθηκε, τι σημαίνει ακριβώς στρατηγική αυτονομία. Πράγματι, είναι μια έννοια που πρέπει να την καθορίσουμε και αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση, δεν πρόκειται για νομικό όρο. Χρειάζεται λοιπόν έναν πολιτικό ορισμό. Με δεδομένη την τρέχουσα πραγματικότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι οποτεδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να αναλάβει μια πρωτοβουλία και έχει ε, αποφασίσει να συνάψει μια σχετική συμφωνία με το ΝΑΤΟ και να αξιοποιήσει κάποιες εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι οποτεδήποτε υπάρχει κάποια αντίθετη άποψη, όπως ο κ έχει μια διαφορετική γνώμη και θέλει να μπλοκάρει αυτέ τι δραστηριότητε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί οι αποφάσει λαμβάνονται με ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι χρειάζεται, και έτσι οδηγούμαστε μάλλον σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείω εξαρτημένη από το ΝΑΤΟ. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι αντιθέτω πρέπει να δημιουργήσουμε μια, τις δυνατότητες να έχουμε και τη δική μας αυτόνομη στρατηγική παρέμβαση, το οποίο συμπεριλαμβάνει επίση και μια βιομηχανία που θα παράγει αυτό που θα χρειαζόμαστε γι' αυτό. Πάντως, συμφωνούμε ότι το, η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας θα πρέπει να διευκρινιστεί. Υποστηρίζοντα και ορισμένε παρεμβάσει άλλων συναδέλφων, θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα στον τομέα τη ε, στρατηγική ασφαλεία και τη ε, εξωτερική πολιτική ασφαλεία, για να έχει ουσία η προσπάθειά μα, πρέπει να υιοθετήσουμε τη λήψη αποφάσεων με αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι με μια αυξημένη πλειοψηφία θα αναγκαστεί κάποιο κράτος μέλος να συμμετάσχει σε μια πολεμική σύραξη που δεν το επιθυμεί. Ε, προς Θεού ούτε καν με ομόφωνη απόφαση δεν μπορεί να αναγκαστεί ένα κράτος μέλος να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ούτε υπό την ΚΕΠΑ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όμως πιστεύω ότι για για, με, με, ένα αποκοδομητικό πνεύμα σε τέτοιες πολιτικές αποφάσεις εκείνοι που δεν το επιθυμούν θα μπορούσαν να απόσχουν και να επιλέξουν και να επιτρέψουν σε αυτούς που το επιθυμούν να συνεργαστούν περισσότερο. Επίσης το ζήτημα της ε, εθνικής κυριαρχίας sovereignty που, που αναφέρεται πολύ συχνά ε, σε ορισμένε περιπτώσει οδηγεί στο να μην έχει κανεί τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Σε ορισμένε περιπτώσει, εάν κάποιο προσπαθήσει με την εθνική του σημαία να παρέμβει, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Επομένω, η εθνική κυριαρχία δεν σημαίνει απλώ το δικαίωμα τη λήψη τη απόφαση, αλλά και τη δυνατότητα επιβολή τη. Εάν οι συνθήκε μας οδηγούν στο να πρέπει να συνεργαστούμε για να υπάρχει όποια πιθανότητα να επιβάλλουμε την απόφασή μας, προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Και για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, η άποψή μα είναι ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε στη λήψη αποφάσεων με αυξημένη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μιχελ Γκάλερ, κυρία Μιχελ Γκάλερ. Τσάρλι Φάιμερ έχει επίση ζητήσει το λόγο. Σικόρσκι. Ο Τσάρλι πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα στην παρέμβαση του κυρίου Γκάλερ για την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο μόνος τρόπος για να έχει κανείς και να διασφαλίσει κανείς την εθνική του κυριαρχία είναι να μην μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες του κράτους στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν δυνατότητες διακυβερνητικών συνεργασιών, συνεργασιών μεταξύ κρατών. Εξάλλου κάτι τέτοιο έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ε, στην Γερμανία και στη Σουηδία, στον τομέα της άμυνας, ακολουθήθηκαν πολιτικές αφοπλισμού, οι οποίες ήταν πολύ καταστροφικές. Ίσως καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν από τέτοιες καταστάσεις, πριν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μεταφέρουμε όλες τις εθνικές αρμοδιότητες των κρατών μέλων στις Βρυξέλλες. Μια και μιλούμε λοιπόν για την της ε, λήψη αποφάσεων με ο, αυξημένη πλειοψηφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιες μικρές χώρες εύκολα θα μπορεί κανείς να τις παραγνωρίσει, να τις πετάξει στην άκρη. Χαίρομαι πάντως που δώσατε και κάποιες ευκρινήσεις, ελπίζω αυτές να συμπεριληφθούν και στην έκθεση. Το είπατε κι εσείς, πρέπει να διευκρινίζετε στην έκθεση τι εννοούμε στρατηγική αυτονομία. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει διεθνή προσωπικότητα, ότι θα μπορεί να λειτουργεί και να δημιουργεί ε, δομές για την ασφάλειά της παράλληλα προς το ΝΑΤΟ. Πρέπει να τα εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε τι εννοούμε εδώ. Ε, διαφορετικά αυτή η συζήτηση δημιουργεί μεγάλη, μεγάλη ανησυχία. Επίση όλοι γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή τη ΚΕΠΑ είναι μια αρμοδιότητα συντρέχουσα μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Μάλλον αυτό είναι η πρόταση. Πώ θα λειτουργεί όμω αυτό. Ε, θα μας ζητούν εθνικές συνεισφορές, θα υπάρχει η δυνατότητα επιβολής ε, από τις Βρυξέλλες ε, στρατολόγησης. Πώς θα λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Γιατί διαφορετικά αν δεν τα εξηγούμε δημιουργούμε ανησυχίες στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριος Να απαντήσω στους συναδέλφους οι οποίοι με ειλικρίνεια υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία. Να τους υπενθυμίσω ότι το δεκαετία του 30 υπήρχε μια απόλυτη εθνική κυριαρχία ε, στις στρατιωτικές αποφάσεις και δεν μας βγήκε σε καλό. Και δεν είμαι σίγουρος αν θέλουμε να το επαναλάβουμε. Για παράδειγμα, η δικιά μου χώρα. Ας πούμε, Πολωνία. Έχει εθνικά συμφέροντα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί και σε άλλες χώρες που ενδιαφέρουν τη Γαλλία. Όχι. Και ποτέ δεν θα στέλναμε στρατεύματα από την Πολωνία σε αυτές τις χώρες, όπως συνέβη στο πλαίσιο ευρωπαϊκών αποστολών, εάν δεν θεωρούσαμε ότι όλοι μαζί αποτελούμε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και άλλα όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να προασπίσουμε κάποιες αξίες που θεωρούμε ότι είναι κοινέ μας. Επομένως, εάν αυτό εννοείται όταν λέτε εθνική κυριαρχία, τότε ανάποδα μην περιμένετε και από εμά να σας βοηθάμε. Επίσης, να επενθυμίσω στους εισηγητές ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια νομίζω έχουμε συμφωνήσει στο συμπέρασμα ότι αυτή η έννοια των ευρωπαϊκών ε, θεάτρων πολέμου ε, περιοχών συγκρούσεων έχει αποτύχει γιατί υπήρξαν τόσο ευρωπαϊκών δυνάμεων έχει αποτύχει γιατί υπήρξαν τόσες επίγουσες καταστάσεις που δεν μπορώ, καταφέραμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε να δημιουργηθούν κάποιες δυνάμεις οι οποίες να μην είναι ε, αποκλειστικά μια σύνθεση εθνικών ε, δυνάμεων. Ε, οι οποίες να μην αποτελούνται από στρατιωτικές μονάδες των κρατών μελών, όπως μέχρι τώρα, αλλά να δέχονται εθελοντές από τα κράτη-μέλη να βρίσκονται υπό πολιτικό έλεγχο του Συμβουλίου και να συντονίζονται και χρηματοδοτικά από την Επιτροπή. Αν δημιουργεί το κάτι τέτοιο ως δύναμη, να δούμε εάν σε κάποια συγκεκριμένη εκπήγουσα στρατιωτική κατάσταση στο μέλλον θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο από τον Ζερόμ και θα σταματήσουμε. Ναι, μια, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, απάντηση. Με εκπλήσει λίγο ε, το, η παρατήρηση που ετέθη σχετικά με μη συμμετοχή σε κεντροαφρικανικές χώρες από ε, συγκεκριμένα κράτη-μέλη, γιατί φαίνεται σαν κατηγορία νεοαπικιοκρατίας ή τέτοιες πολιτικής ε, προς τη χώρα μας θυμίζω στον αγαπητό συνάδελφο ότι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαθα εκεί είναι για να μην φτάσει η Ισλαμική τρομοκρατία στο έδαφος μας, εδώ στην Ευρώπη. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η ασφάλεια όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, εκεί όπου διαχέονται ανοιχτά ιδέες ε, των Ισλαμικών ε, τρομοκρατικών ομάδων, μάλλον είναι μια σημαντική αποστολή. Ωραία, πιστεύω ότι θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Ξέρω ότι ο ε, ε ανυπομονεί και για τη δική του ε, συνάντηση ε, των σκιωδών, όσο περιμένω και εγώ τη δικιά μου. Θα, τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Τώρα για τα διάφορα δεν έχουμε κάτι. Οι επόμενες συναντήσεις, η αφέτε ε, θα κάνει ε, μια έκτακτη συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου των, ε, στις Βρυξέλλες στην συνέχεια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤΣΕΝΤ στις 21 Νοεμβρίου 11.30 με 1 για ανταλλαγή απόψεων με τον Ζαμπιέρ Λακουά αντικαθιστά την Γενική Διευθύντη του ΟΗΕ για δράσεις για την ειρήνη, ενώ στο Στρασβούργο την επόμενη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ ΝΤΕΒΕ Ντρουά για ανταλλαγή απόψεων με τον Άλεξ Σετσόφ, ο οποίος έλαβε το ε, βραβείο Σακχάροφ για το 2018. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της ε, συνεδρίασης και παρακαλώ τους ε, συντονιστές των παρατάξεων να ε, παραμείνουν ε, στην αίθουσα. Ε, φυσικά και όλες οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να μείνουν, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την επιστολή μας. Εδώ λίγη συνεδρίασή μας. Ευχαριστούμε τους αντιπροσώπους από την Γεωργία και θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά.